που έχει υποβάλει ο κύριο Δανιέλ Κάσπαρη και οι προτάσει αυτέ παραπέμφθηκαν σε αρμόδιε επιτροπέ. Και τώρα περνάμε στην ημερήσια διάταξη. Το οριστικό σχέδιο ημερήσια διάταξη ορίστηκε στι 6 Απριλίου από τη διάσκεψη των Προέδρων σύμφωνα με το άρθρο 149 και έχει διανεμηθεί. Σύμφωνα, μετά μάλλον από διαβουλεύσει με τι πολιτικέ ομάδε, θέλω να υποβάλω στην Σύνοδο την εξή πρώτα τροποποίηση τη οριστική ημερήσια διάταξη για την Τετάρτη ε, η σειρά του δεύτερου και του τρίτου σημείου αντιστρέφονται, ούτω ώστε η δήλωση της Επιτροπής για την απόφαση που εθετήθηκε σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, με την πρωτοβουλία για την ε, ε, ισορροπία μεταξύ εργασιακή και προσωπικής ζωής, θα είναι δεύτερο σημείο μετά από τη δήλωση της Επιτροπής για την Ουγγαρία. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, εγκρίνεται και τροποποιείται έτσι η ημερήσια διάταξη. Επιπλέον, Κύριε Πιτέλα, παρακαλώ. Όχι για αυτό που μόλις είπατε, γι' αυτό συμφωνούμε. Αλλά θα ήθελα να προτείνω μετά από τη συζήτηση που θα γίνει για την Ουγγαρία να προβλέψουμε και σχετικό ψήφισμα για τον Μάιο. Όπως είπε ο κύριος Σπιτέλα, ε, ζήτησαν, ε, η ομάδα των σοσιαλιστών ζήτησε μετά από τη συζήτηση για την κατάσταση στην Ουγγαρία να υπάρξει ψήφισμα το οποίο θα ψηφιστεί την πρώτη σύνοδο του Μαΐου. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Πιτέλα για να ε, παρουσιάσει αυτή την πρόταση. Όχι, το έκανε ήδη, τέλεια. Υπάρχει κάποιος που είναι αντίθετος με αυτό το αίτημα του κύριου Πιτέλα. Είστε κατά. Υπάρχει κάποιος που είναι κατά της πρότασης του κυρίου Πιτέλα. Ο κύριος Γιούρικ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ευρώπη είχε πολλές συγκρούσεις ε, μέχρι τώρα. Δεν χρειάζεται να αρχίσουμε άλλη μια σύγκρουση με μια χώρα που απλώς θέλει να έχει τη δικιά της πολιτιστική πολιτική. Μπορούμε να το κάνουμε αν το επιθυμεί αυτό το Κοινοβούλιο, να ξεκινήσουμε ψήφισμα και σύγκρουση με μία παραπάνω χώρα νομίζω ότι μας βάζει ακόμα πιο βαθιά στην κρίση. Κανείς δεν νιώθει αλληλεγγύη με την Ουγγαρία, αλλά ανεξάρτητα με τις δικές μας πεπιθήσεις δεν πρέπει να βάλουμε πιο βαθιά στην κρίση την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Μάλιστα τότε θα ψηφίσουμε. Ναι, παρακαλώ. Η κυρία Βεριζιά, για διαδικαστικό. Κύριε Πρόεδρε, μια διευκρίνηση για το αίτημα του κυρίου Πιτέλα. Υπήρχε συμφωνία μεταξύ διάφορων πολιτικών ομάδων ούτω ώστε να υπάρξει και αίτημα ψηφίσματος και αίτημα αποστολής στην Ουγγαρία. Θα ήθελα η πρόταση αυτή να τεθεί σε ψηφοφορία από κοινού, τα δύο τη δηλαδή, όπως είχαμε συμφωνήσει. Κυρία μου, εγώ έλαβα το αίτημα του κυρίου Πιτέλα εξ ονόματος ε, ε, ε, της Σοσιαλιστική Ομάδας του Κοινοβουλίου μετά τη συζήτηση να υπάρξει ψήφισμα το οποίο θα ψηφιστεί τον Μάιο. Δεν υπευλήθη αίτημα για διοργάνωση κάποια αποστολή. Quindi mi pare che la si pronuncia su Οπότε εμείς μπορούμε ω Σύνοδος να αποφασίσουμε μόνο για την ημερήσια διάταξη. Δεν υπάρχει λοιπόν κάποιο τέτοιο αίτημα, οπότε θα ψηφίσουμε για την πρόταση του κυρίου Πιτέλα και των σοσιαλιστών για ψήφισμα για την κατάσταση στην Ουγγαρία που θα ψηφιστεί στη σύνοδο, την πρώτη σύνοδο του Μαΐου. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Οπότε, η συζήτηση επί της δήλωσης της Επιτροπής για την κατάσταση στην Ουγγαρία θα ολοκληρωθεί με ψήφισμα το οποίο θα ψηφιστεί στην πρώτη σύνοδο του Μαΐου. Έλαβα επίσης το εξής αίτημα. Η Ομάδα Ευρώπη των Εθνών και της Ελευθερίας ζήτησε ε, ότι η δήλωση, τη δήλωση ε, του Αντιπροέδρου της Επιτροπής είπα της εκπροσώπου ε, να προσθεθεί μετά από τη συζήτηση για τη Συρία μία συζήτηση για τη συγκατάσταση των κοπτών στην Αίγυπτο και η συζήτηση για την έκθεση του κυρίου Διακόνου για το έτος της πολιτιστικής κληρονομιάς να αναβληθεί για τον Μάρτιο. Εδώ δίνω το λόγο στον κύριο Μπερμάγερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στις 9 ε, Απριλίου, την Κυριακή των Βαΐων, έγιναν τρομοκρατικές ε, επιθέσεις κατά των ε, χριστιανών κοπτών στην Αίγυπτο, όπου βρήκαν το θάνατο 78 κόπτες. Είναι το τελευταίο επεισόδιο της τεράστιας τρομοκρατικής εκστρατείας κατά των 10 εκατομμυρίων κοπτών της Αιγύπτου. Με βάση το άρθρο 149α Θέλω να θέσω αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη και σας παρακαλώ να μας υποστηρίξετε και να υπάρξει ονομαστική ψηφοφορία γι' αυτό. Και πρέπει να θυμηθούμε ότι και ο Πάπας ε, Φραγκίσκος ε, ε, ετοιμάζεται να υποστηρίξει και ενδεχομένως και μεταξύδι τους κόπτες. Ευχαριστούμε κύριε Ομπερμάγερ. Θέλει κανείς να μιλήσει κατά. Κατά. Ο κύριος Πρέδα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συζήτηση για τους χριστιανούς σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Είναι καλό να κάνουμε τέτοια συζήτηση το Μάιο. Τώρα, αύριο ξέρετε ότι θα συνεχθείτε με το μεγάλο μουφτή της Αιγύπτου και σίγουρα θα του εκφράσετε τις ανησυχίες μας για την κατάσταση των κοπτών. Τη συζήτηση για τους χριστιανούς να την κάνουμε τον Μάιο πάντως, γιατί η σε διάταξη είναι ήδη πολύ φορτωμένη. Κύριε Ομπερμάγερ, επιμένετε σε αυτή σας την πρόταση για συζήτηση για την κατάσταση των κοπτών στην Αίγυπτο σε τούτη εδώ την σύνοδο ή μήπως ε, προτιμάτε την πρόταση του κυρίου Πρέντα ώστε να γίνει η συζήτηση τον Μάιο και έπειτα βέβαια η διάσκεψη των Προέδρων θα το συζητήσει. Κοιτάξτε, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα οξία. Δεν μπορούμε να το αναβάλουμε. Υπάρχουν πολλά θέματα που επίσης είναι ιδιαίτερα οξυμένα και θεωρώ ότι πρέπει να το θέσουμε στη μέρη διάταξη. Πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Να το θέσουμε στη μέρη διάταξη. Σχετίζεται ακριβώ και με την επίσκεψη που είπα του Πάπα Φραγκίσκου στην Αίγυπτο. Πρόεδρε, να σας ενημερώσω τι θα γίνει τώρα. Υπάρχουν δύο προτάσεις που έχουμε. Υπάρχει πρόταση του κύριου Πρέντα που πρέπει να ψηφιστεί, γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό να το ξέρουμε. Παρόλο που έχω κάθε συμπάθεια για την ε, πρόταση Μπερμάγερ, υπάρχει και η δεύτερη όμως πρόταση, την οποία νομίζω ότι πρέπει να ψηφίσουμε τώρα. Και ως η πρόεδρος της σχετικής διακοινοβουλευτικής ε, ε, ομάδας θα ήθελα να ψηφιστεί η πρόταση Πρέντα για να ξέρω τελικά. Μπορείτε να μας πείτε τι ψηφίζουμε ακριβώς. Ο κύριος Μποστινάρο. Πρόεδρε, συμφωνώ απόλυτα με την ιδέα του να συζητήσουμε την κατάσταση αυτή, αλλά πρώτον, ποιο να κατηγορήσουμε, γιατί η κυβέρνηση, οι αρχές, το κράτος κάνουν ό,τι μπορούν για να αποφύγουν τρομοκρατικές ενέργειες. Οι τρομοκράτες είναι τρομοκράτες και τα θύματα είναι θύματα. Αυτό είναι το μόνο που γνωρίζουμε. Και δεν είναι θέμα να συζητήσουμε την θρησκευτική διάσταση σε αυτά. Γι' αυτό δεν μου αρέσει η ιδέα του να στοχεύσουμε μια συγκεκριμένη ομάδα και να μην δώσουμε υπερβολική διάσταση στην θρησκευτική πτυχή της τραγωδίας αυτής. Λάουλα Σοβράνα. Το... Εσείς αποφασίζετε, η Ολομέλη αποφασίζει. Λοιπόν, ψηφίζουμε για το αίτημα της Ομάδας Ευρώπη των Εθνών και της Ελευθερίας ε, ε, που υπέβαλε ο κύριος Σόμπερ για να προσθέσουμε στην ημερήσια διάταξη αυτή εδώ τη Συνόδου μετά από τη συζήτηση για την Τουρκία μια συζήτηση με δήλωση της ΥΠΑ της εκπροσώπου για την κατάσταση των κοπτών στην Αίγυπτο. Η ε, ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε τη ψηφοφορία. Η πρόταση απορρίπτεται. Όσον αφορά το αίτημα του κυρίου Πρέντα, όπου νομίζω πως υπάρχει, μάλιστα, παρακαλώ, η κυρία, η κυρία Μπερές. Δεν θα αλλάξει το αποτέλεσμα, αλλά θέλ, ήθελα να σας πω ότι δεν έχω την κάρτα μου και θα καταψήφιζα. Allora, vi propongo... Οπότε, σας προτείνω την εξής λύση. Καθώς η διάσκεψη των Προέδρων αποφασίζει για την ημερήσια διάταξη της Συνόδου του Μαΐου, υπαριθμόν 1, θα πρέπει να μπει στην ημερήσια διάταξη της σκέψης των Πρόεδρων το αίτημα του κυρίου Πρέντα που υποστηρίζεται και από τους σοσιαλιστές όπως φάνηκε από τα όσα είπε ο κύριος Μπουστινάρο οπότε δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε τώρα γιατί στη συνέχεια η διάσκεψη των Προέδρων θα αποφασίσει πάντως νομίζω πως υπάρχει πλειοψηφίο, να συζητηθεί στην πρώτη σύνοδο του Μαΐου το θέμα της κατάστασης των χριστιανών στον κόσμο ε, γενικότερα θα αναλάβω αύριο ε, στην συνάντησή μου με τον ε, Μέγα Μουφτή να υπογραμμίσω πόσο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σημαντική η ανοχή, ο διάλογος ανάμεσα στις θρησκείες και η συμβίωση ε, ανάμεσα στις διάφορες θρησκείες. Γιατί στην Αίγυπτο η πλειοψηφία είναι μουσουλμάνοι, αλλά υπάρχουν και γύρω στα 10 εκατομμύρια χριστιανοί και άρα και η προστασία των μειονοτήτων είναι σημαντική για μας, όπως κάνουμε άλλωστε και εμείς στην Ευρώπη αυτό το μήνυμα θα το παραδώσω άμεσα στον ε, μεγάλο μουφτή, τον οποίο θα συναντήσω αύριο εδώ στην έδρα του Ευρωκοινοβουλίου. Και στη συνέχεια η διάσκεψη των Προέδρων θα επικυρώσει αυτή την απόφαση που νομίζω μας βρίσκει σύμφωνος. Να σας ενημερώσω εξάλλου ότι την Πέμπτη η Νομική Επιτροπή ενέκρινε την εξή έκθεση για την ε, ασυλία του κυρίου Λεμπρετών. Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 8 του κανονισμού του Κοινοβουλίου η έκθεση αυτή θα ψηφιστεί την Πέμπτη. Στην ώρα της ψηφοφορίας, επιπλέον η ΓΚΟΕ έχει υποβάλει σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφο 3 του κανονισμού του Κοινοβουλίου μια πρόταση ε, αντίρρηση στην Κομισιόν ε, και στον προτινόμενο κανονισμό που τροποποιεί το παράρτημα 2 του κανονισμού 978-2012 και που εφαρμόζει ένα σύστημα γενικευμένων ε, δασμολογικών προτιμήσεων. Αυτό θα ψηφιστεί και αυτό στη διάρκεια τη ώρας των ψηφοφοριών την Πέμπτη και έτσι θα έχει η ημερήσια διάταξη με αυτές τις ε, μικρές αλλαγές. Και τώρα θα περάσουμε στην δήλωση της Επιτροπής για την κατάσταση στην Ουγγαρία. Το λόγο έχει ο πρώτος αντιπρόεδρος, κύριος Φραντς Τίμερμανς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη, κύριε Πρωθυπουργέ. Οι πρόσφατες εξελίξεις στην Ουγγαρία έχουν προκαλέσει πολλές ανησυχίες σε πολλά άτομα και στην Ένωση και ευρύτερα. Συμμεριζόμεθα αυτές τις ανησυχίες.